να μην ε, σβήσει τελείω από το μέλλον. Εάν η Τουρκία ε, πληρώσει προποθέσει, να μπει. Εάν όχι, όχι. Ο καθένα από εμά όμω θα πρέπει να ε, αναζητήσει του κατάλληλου μηχανισμού που να προωθούν και να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και και τη δημοκρατία σε τρίτε χώρε. Γι' αυτό πρέπει να υποστηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών. Αυτό είναι πρώτη τη σημασία. Ευχαριστούμε και για την λάθος προφορά του ονόματός σας, να με συγχωρείτε. Ε, κυρία Ροντρίγκς. Τώρα, συνάδελφοι, προχωράμε στη διαδικασία ΚΑΤΣΤΙΑΕ. Uh, Θα παρακαλέσω τους συμμετέχοντες να παραμείνουν αυστηρός στο ένα λεπτό. Ο κύριος Λίντς. Συγχαρητήρια στην Κάτι για την ε, πολύ καλή έκθεση για την ε, κατάσταση του ΚΙΑ που γίνεται όλο και πιο δραματική. Έχουμε ε, πάνω από 10.000 κρατήσεις, προσαγωγές συνεχώς. Η Ρεμπέκα Χάρμς έχουμε παρακολουθήσει δίκες. Ο δημοσιογράφος Ντουντάρ Ξέρουμε ότι διώκεται η σύζυγός του, δεν έχει πλέον διαβατήριο. Έχουμε Γερμανούς δημοσιογράφους ε, που δεν έχουν πλέον διαπίστευση ε, και από το Τσεντεφ και από το Τάγκε Σπίγκελ. Δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους πλέον. Αυτά τα καταδικάζουμε περίφραστα και δείχνουν πόσο πλήττεται η ελευθεροτυπία στην Τουρκία. Γι' αυτό είναι σημαντικό Επίσημώ ε, να ζητήσουμε την αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Όμω ε, δεν είμαστε υπέρ της ε, πλήρους παύσης, της διακοπής του οριστικής, διότι δεν θέλουμε να πλήξουμε την κοινωνία των πολιτών. Θέλουμε να μπει στο δρόμο τη δημοκρατία χώρα. Ευχαριστώ κυρία Ward be in Turkey since the beginning of my mandate. να στην Τουρκία ε, και τη πράσπιση του δημοκρατικού Και είναι πολύ ε, ατυχέ πόσο άσχημα έχουν πάει τα πράγματα τα τελευταία πέντε χρόνια. Η σύσταση για την αναστολή των ε, ενταξιακών διαπραγματεύσεων είναι δυστυχώ οδυνηρό μήνυμα, διότι η Τουρκία θα χάσει την πορεία τη προ την Ευρώπη. Επαφέ με την κοινωνία των πολιτών με πείθει ότι λαχταράνε για δημοκρατική πρόοδο και ανθρώπινα δικαιώματα οι πολίτε στην Τουρκία. Όμω οι διώξει των συνδικαλιστών, ακαδημαϊκών, ε, πανεπιστημιακών, των εθνοτικών μειονοτήτων, των ΛΟΑΔ, κάνει αδύνατο να συνεχίσουμε έναν διάλογο που να φέρεται επικοδομητικό. Ο κύριο, ε, η κυρία ε, Εντόαν, η οποία ήταν φεμινίστρια και καλλιτέχνη, συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα τη Human Rights Watch για την προστασία των δημοσιογράφων, πρόσφατα απελευθερώθηκε. Όμω η υπόθεσή τη δείχνει πώ ακριβώ οι τουρκικέ αρχέ μπορεί να στοχεύσουν οποιονδήποτε ασκεί και εναντίον του. Η απεργία πείνα εκατοντάδων ε, Κούρδων αυτή τη στιγμή, γιατί έχει μπει στην απομόνωση η Αβδέλα Ζουλάν, δείχνει ότι υπάρχει τεράστια δυσαρέσκεια κατά του καθεστώτο του Ερντογάν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριο Μαυρίδη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τι είναι σήμερα η Τουρκία, μια ανοιχτή φυλακή με μαζική παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατάλυση του κράτους δικαίου έξω από την τουρκία μια επεκτατική δύναμη που παραβιάζει το διεθνέ δίκαιο και με ισλαμιστική πολιτική ατζέντα. η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε δυστυχώ δηλητηριασμένη με τα οικονομικά συμφέροντα και τι πολιτικέ επιδιώξει επιμέρου κρατών ει βάρο των αξιών μα, το πιο τρανό παράδειγμα οι υποχρεώσει τη Τουρκία προ την ευρωπαϊκή ένωση που αφορούν ένα μικρό κρατο μέλος την κυπριακή δημοκρατία ουδέποτε εκπληρώθηκαν. παρεμπιπτόντως τέτοια πολιτική υποκριτική από την ευρωπαϊκή ένωση τροφοδοτεί τις αντιευρωπαϊκές δυνάμεις οι οποίες θέλουν να καταστρέψουν το ευρωπαϊκό εγχείρημα. για να έχουμε λοιπόν αξιοπιστία η πολιτική επιβολής κυρώσεων και εμπάρκο πώλησης όπλων έπρεπε να είναι ήδη στην έκθεση. λυπάμαι που δεν είναι μέσα και πολύ περισσότερο λυπάμαι γιατί δυστυχώς κάποιοι θα το έχετε μετανιώσει στο μέλλον. Ευχαριστούμε κυρία Μιράντα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Ερντογάν έχει καταστρέψει τι κρατικέ αρχέ και του φορεί τη Τουρκία. Αυτό φαίνεται ιδίω με τη δίωξη κατά την καταστολή κατά των ε, αντιφρονούντων. Και αυτό κυρίω κατά των Κούρδων και του, ΧΑΝΤΕΠΕ. Ο ε, κύριος κύριο Ερντογάν ε, έχει βάλει στην φυλακή τον κύριο Δημαρτά και εγώ πήρα υποστολή από εκείνον που λέει ε, από τον Δεκέμβριο ότι ζητάει να παγώσουν οι διαπραγματεύσει με την Τουρκία. Όχι απλώ να σταλούν, να πάυσουν. Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει το διάλογο, κύριε Επίτροπε, τον διαφανή διάλογο με την Τουρκία, ασκώντα κριτική κατά των κακώ προπραγμένων τη Τουρκία, να απαιτήσει τοπικέ εκλογέ. Αλλά ε, η Τουρκία και ο κουρδικό και τουρκικό λαό δικαιούνται τη συνεργασία και τη στήριξή μα. Μην του αφήσουμε στην τύχη του στα χέρια των δικτατόρων. Δικτατόρων που φυλακίσαν περισσότερου από 50.000 δημοσίου υπαλλήλου. Περισσότερου από 2.000 κυβερνητικέ οργανώσει τι κλείσανε και 200 μέσα μαζική ενημέρωση και βουλευτέ. Συγγνώμη, αλλά τέλειωσε η ώρα σα. Ο κύριο Ηλικιώτη, για ένα λεπτό. Η Τουρκία συνεχίζει την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών του λαού τη, ενώ κατέχει παράνομα και δια της βίας των όπλων εδάφιους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απαράδεκτο να ζητείτε αναβάθμιση τη Τελωνιακής Ένωση όταν η τουρκία αρνείται να εκπληρώσει πλήρω και χωρί διακρίσει τι υποχρεώσει που απορρέουν από την τρέχουσα συμφωνία και αρνείται να αναγνωρίσει την κυπριακή δημοκρατία. το ελκ σε μια επίδειξη λαϊκισμού προτείνει τον τερματισμό των ενταξιακών διαπραγματεύσεων την ίδια ώρα που τάσσεται υπέρ τη άνευ προποθέσεων αναβάθμιση τη τελωνειακή ένωση. σα καλούμε συνάδελφοι να καταψηφίσετε την πρόταση για άνευ προποθέσεων αναβάθμιση τη ένωση καθώς αντιβαίνει κάθε κανόνα λειτουργίας της ένωσης και κάθε έννοιας δικαίου. την ίδια στιγμή αναμένουμε από την ένωση να ασκήσει πιέσει προς την τουρκία ώστε να υλοποιήσει όλες τις κυπρογενείς της υποχρεώσεις να τερματίσει τις παράνομες ενέργειες στην κυπριακή ΑΟΣ. να αποσύρει τον κατοχικό στρατό από την κύπρο να τερματίσει τον επικισμό και να συμβάλλει έμπρακτα στην επίλυση του κυπριακού στη βάση τη ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία όπω καθορίζεται στα ψηφίσματα του συμβουλίου ασφαλεία του οηε. ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή στη φωτογραφία είναι η Λαγούβαν από τις 8 Νοεμβρίου σε απεργία πείνας. Ε, απεργία πείνας για να ζητήσει μεταξύ άλλων να βγει από την απομόνωση ο Τσαλάν ε, έχει μείνει 20 χρόνια στις φυλακές της Τουρκίας σε απομόνωση. Στην Τουρκία βλέπουμε μια κατάσταση έκτατης ανάγκης που έχει γίνει μόνιμη μετά την απόπειρα προξυποκοπήματος που ουσιαστικά ε, χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα για να παγιωθεί ένα πολιταρχικό καθεστώς. Εγώ πήγα ίδια στην Άγκυρα για να προσπαθήσω να παραστώ στη δίκη των δύο προέδρων του ΚΑΝΤΕΠΗ, του ΧΑΝΤΕΠΕ που ήταν ε, ε, στα χέρια της δικαιοσύνης, όπως του Ντεμέρ και μαζί και του Ντεμέρτα, του... αλλά δεν μου δόθηκε δικαίωμα πρόσβασης. Θα... Και εγώ προσπάθησα, θα προσπαθήσω να χαιρετήσω τα άτομα που βρίσκονται εδώ στο Στρασβούργο σε απεργία πείνα σε αλληλεγγύη προ την ε, Λαγούβαν για να βγει ο Τσαλάν από την απομόνωση στι φυλακέ. Θα πρέπει να τοποθετηθεί και για αυτό το Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστούμε κύριο Φουντούλη για ένα λεπτό τελευταίο. Η Τουρκία ακόμα και γεωγραφικά δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα δεν ασπάζεται και δεν επιθυμεί να ασπαστεί τι αξίε του δυτικού πολιτισμού κάνει διακρίσει ει βάρο των θρησκευτικών μειονοτήτων συμπεριλαμβανομένων των χριστιανών και των αλεβιτών. η κυβέρνηση ερντογάν καθημερινά απολύει και διώκει δημόσιου υπαλλήλου δασκάλου γιατρού ακαδημαϊκού δικηγόρου δικαστέ και εισαγγελεί. η τουρκία με εισβολή από το 1974 κατέχει παράνομα μεγάλο τμήμα τη κύπρου. η τουρκία ακολουθεί επιθετική πολιτική εναντίον τη ελλάδο παραβιάζει καθημερινά τον εναέριο χώρο και τα χωρικά ύδατά τη αρνείται να υπογράψει και να ακυρώσει τη σύμβαση των ηνωμένων εθνών για το δίκαιο της θάλασσα. η τουρκία υποστηρίζει και χρηματοδοτεί την τρομοκρατία. απαιτούμε την άμεση επίσημη και οριστική διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων απαιτούμε την πλήρη διακοπή κάθε ευρωπαϊκής οικονομικής ενισχύσεως προς την τουρκία και επιπλέον την εφαρμογή οικονομικών και άλλων κυρώσεων. ζητάμε την επίσημη αποκήρυξη εκ μέρους τουρκίας κάθε επεκτατική διεκδικήσεως εις βάρος της ελλάδος και την πλήρη και ανεφόρον απελευθέρωση των κατεχομένων τη κύπρου. μέχρι τότε αυτό το κράτο δολοφόνο δεν έχει καμία θέση στο ίδιο τραπέζι με τα κράτη μέλη τη ενώσεως. στην ευρωπαϊκή ένωση η τουρκία ούτε έχει και ούτε θα πρέπει να έχει ποτέ θέση. ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε. Ο Πίτροπος Χάν παρακαλώ τώρα να κάνει κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι σας ευχαριστώ όλες και όλους για τις παρεμβάσεις σας, για τις παρατηρήσεις σας. Νομίζω ότι όλοι ανισχούμε εξίσου με την κατάσταση των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας ε, και ε, Εμεί ε, έχουμε ήδη πει, όπως είπε το Συμβούλιο, ότι ήδη υπάρχει αυτή τη στιγμή αναστολή, πάγωμα ε, των διαπραγματεύσεων ε, με την Τουρκία. Ε, το θέμα είναι όμως να παραμείνουν κάποιοι διάβλοι ανοιχτοί με την Τουρκία και Ξέρω ότι δεν συμφωνούν όλοι με αυτό, αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι ε, η αναβάθμιση της τελωνιακής σχέσης ε, ένας ε, τρόπος να ανοίξει και πάλι ένας διάβλος επικοινωνίας. Φυσικά και η Τουρκία θα πρέπει να σέβεται τους κανόνες της συμβάσης που έχει υπογράψει και ως υποψήφια χώρα, ως μέλος επίσης του Βουλού της Ευρώπης και υπογραμμίζουμε την ανάγκη Άγκυρα να κάνει βήματα ξεκάθαρα για τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπινών δικαιωμάτων και να διορθώσει τα επίμαχα διμερεί προβλήματα ε, με τις ε, γειτονικέ της χώρες. Θα συνεχίζουμε να εμένουμε σε αυτό και σε ό,τι αφορά το ετήσιο πακέτο διεύρυνσης ε, την Άνοιξη θα αναφέρουμε ε, τις απόψεις μας για μια ακόμη φορά. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και Πρέπει να πω ότι η δημοκρατική κοινωνία ξεκινά με θεσμικά αντίβαρα, ξεκινά με λογοδοσία. Ευχαριστώ και τώρα η κυρία Υπουργό Τσιότ έχει το λόγο. Honorable members, and Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω κατά κλείδι να ευχαριστήσω για την χρήσιμη συζήτηση. Άκουσα προσεκτικά τις απόψεις σας και σημειώνω ότι και η δική μας εκτίμηση είναι παρόμοια σε πολλά θέματα προσβλέπουμε στη συνέχιση του δημιουργικού διαλόγου. Σας διαβεβαιώνω ότι το Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Τουρκία. Προσέχοντας ιδιαίτερα τα θέματα που συζητήσαμε σήμερα εδώ. Η προσεχής 54η Σύνοδος του Συμβουλίου Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας την Παρασκευή 15 Μαρτίου θα αποτελέσει μια εξαιρετική ευκαιρία όχι μόνο ανασκόπηση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, αλλά και μια ευκαιρία συζήτησης των προκλήσεων και των ευκαιριών που έχουμε μπροστά μας. Θα μεταφέρω στους Τουρκου συνομιλητές μας το απερίφραστο μήνυμα, το ομόφωνο μήνυμα, ότι πρέπει χωρίς καθυστέρηση να αντιμετωπίσουν τα θέματα που εντοπίσετε κι εσείς στη σημερινή σας έκθεση, ε, όπως και τις παρατηρήσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Ταυτοχρόνως πιστεύω ότι όλοι έχουμε να κερδίσουμε αν εντείνουμε τον διάλογο με την Τουρκία σε όλα τα επίπεδα. Από την πλευρά μας, από την πλευρά της Προεδρίας, μαζί με τα κράτη-μέλη και την Κομισιόν, θα συνεχίσουμε να πράττουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Εν τέλει, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συμβολή του και για τις προσπάθειες της εισηγήτριας Κάτι Πύρη που προέβη σε μια συνολική επισκόπηση των εξελίξεων στην Τουρκία. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σημαντικός στην ευρύτερη διαδικασία εντός της οποίας δρούμε και εμείς. Έτσι δίνουμε την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη διαδικασία οι πολίτε τη Τουρκία αλλά και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. σε δημοκρατικέ δηλαδή ανταλλαγέ απόψεων, κάτι το οποίο είναι προ το συμφέρον τόσο τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τη Τουρκία. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Υπουργό και παρακαλώ την εισαγήτρια κυρία Κάτι Πύρη για δύο λεπτά για να κλείσει η συζήτηση. Thank you, Commissioner. Ευχαριστώ Επίτροπε Υπουργέ, ευχαριστώ συνάδελφοι. Καταρχάς, να επανέλθω σε αυτό που είπε το Συμβούλιο εκ μέρου τη Προεδρία. Λέτε όλοι οι δίευλοι επικοινωνία πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί. Επικοινωνία με την Τουρκία. Συμφωνούμε όλοι. Όμω ε, ο διάβλο και η οδό τη ένταξη πρέπει να κλείσει. Έχει γίνει γελίο πλέον αυτό. Επίση, λέτε ότι σημειώνουμε και συνεχίζουμε να παρακολουθούμε. Χαίρομαι που στο συμπερασμά σα την Παρασκευή μετά τη συνάντηση με την Πρόεδρο της Τουρκίας είπατε ότι πρώτο τι προτεραιότητά σα θα είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Χαίρομαι για αυτή την υπόσχεση, όμω α μα πει το Συμβούλιο πώ θα βοηθήσει του δημοκράτε τη Τουρκία. Θα του δώσουμε κονδύλια, θα στηρίξουμε του υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα βάλετε το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων ω βασικό κριτήριο για τη συνέχιση των εμπορικών σχέσεων. Πραγματικά ελπίζω το Συμβούλιο να βρει κάτι λίγο πιο συγκεκριμένο στη στρατηγική του για να το πει, αντί για αυτά που ω τώρα έχουμε δει να εφαρμόζονται ε, σε σχέση με την Τουρκία. Και άκουσα το πολύ μάλλον δεν άκουσα ούτε πέντε συναδέλφου να λένε εδώ σε, αυτό το, σε αυτή τη συζήτηση ότι αυτή η και δεν θα έχει καμία ε, επίπτωση στι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Το είπαμε. Να σταματήσουν οι ενταξιακές ε, με σκοπό την προσχώρηση με τον πρόεδρο Ερντοχάν. Δεν έχει καμία λογική. Γίνεται και εξωφρενικό και ανοητό. Επίση, άκουσα να λένε κάποια μέλη τη ακροδεξιά ότι υπάρχουν μέλη του ΕΛΚ που ήθελαν να πάνε ένα βήμα παραπέρα. Ε, να ε, μην έχει πια κάνει το καθεστώ υποψήφια χώρα στην Τουρκία και αυτό να το ε, υποστηρίξουμε. Ε, Εκπλήσω που το ακούω αυτό, γιατί επί 10 χρόνια είχαμε εισηγητή του ΕΛΚ που ποτέ δεν έκανε τέτοια έκκληση. Εάν πραγματικά μιλάτε για παραβιάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τότε ακολουθήστε αυτό που λέει η πλειοψηφία του σώματο αυτού του Κοινοβουλίου. Ε, διότι ζητήσαμε αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και ελπίζω τα επόμενα χρόνια, τι ερχόμενε δεκαετίε, η Τουρκία να μπορέσει να βελτιωθεί. Ελπίζω ότι όλοι ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή στο εσωτερικό τη Τουρκία τα πράγματα μπορεί και να αλλάξουν και ε, θα δούμε αν είναι οριστικό και για πάντα το τέλο των ενταξιών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε, συνάδελφε. Έληξε η συζήτηση. Αύριο θα γίνει η ψηφοφορία. Και τώρα μια-δυο ανακοινώσει. Χθε ο πρόεδρο ανακοίνωσε ότι το άρθρο 171 εδάφιο 1 σημείο β του ιστορικού κανονισμού ε, όπω το πρότεινε η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων στην ερμηνεία του, εγκρίνεται. Αν δεν υπάρξουν άλλε αντιρρήσει μέσα σε ένα 24ωρο, η ερμηνεία αυτή του άρθρου θα εγκριθεί βάσει του άρθρου 226. Επόμενη ανακοίνωση για τις συστάσεις περί αποφάσεων από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων να μην υπάρξουν αντιρρήσεις για τις καταξιότητες πράξεις και την ε, ε, και εφόσον δεν υπήρξαν αντιρρήσει μάλλον για τι κατεξοδοτήσει πράξει μέσα σε 24 24ωρο, βάσει το άρθρο 105 παράγραφο 6, οι συστάσει αυτέ θεωρούνται εγκεκριμένε. Θα εγκριθούν μαζί τα υπόλοιπα εγκεκριμένα κείμενα από αύριο, Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019. Και τώρα, συνάδελφοι, να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, που είναι δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής, είπα της εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, για το θέμα της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα. Βεβαίως, εκ μέρους της είπα της εκπροσώπου θα πάρει το λόγο Επίτροπος. Έχετε το λόγο Επίτροπε. Ε, εδώ καλωσορίζουμε την ε, στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση ανάγκη στην Βενεζουέλα και την έκκλησή σα για να βρεθεί μια μόνιμη λύση στη χώρα. Πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στα διάθεσή μα για να βρούμε μια ειρηνική και δημοκρατική λύση μέσω ελεύθερων και αξιόπιστων προεδρικών εκλογών από την τελευταία μας συζήτηση για τη Βενεζουέλα στην ε, Ολομέλεια αυτή στο τέλος του Ιανουαρίου οι εντάσεις και η πόλωση ε, προχώρησαν. Ε, οι συνθήκες διαβίωσης υποβαθμίστηκαν περαιτέρω. Ο αριθμός των κατοίκων της Βενεζουέλας που εγκαταλείπουν τη χώρα ε, διωγγώνεται. Και βάσει της ΥΠΑ της Αρμοστίας για τους πρόσφυγες του ΟΗΕ, 2,7 εκατομμύρια Βενεζουελάνοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους από το 2015. Ο αριθμός συνεχίζει να αυξάνεται. Μπορεί να φτάσει και τα 5 εκατομμύρια μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς, εάν συνεχιστεί η τωρινή κρίση. Ε, ο το blackout που χτύπησε και έπληξε ολόκληρη τη χώρα και ακόμη συνεχίζεται σε κάποια κράτη της Βενεζουέλας έχει πλήξει την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και την παροχή νερού, την υδροδότηση. Όπως όλοι γνωρίζουμε αυτά τα blackout, αυτές οι βλάβες ε, έχουν την ε, πηγή τους στα πολιτικά και θεσμικά προβλήματα. Η τωρινή κατάσταση έχει προκαλέσει επιθέσεις κατά της δημοκρατίας, του συντάγματος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η λύση στην κρίση θα πρέπει να είναι πολιτικού χαρακτήρα αλλά και δημοκρατικού να είναι ειρηνική και να την έχει ε, βάλει σε πράξη ο ίδιος ο λαός της Βενεζουέλας. Πρέπει να απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι και θα πρέπει να αποκατασταθούν όλα τα δικαιώματα της Εθνοσυνέλευσης. Η Εθνοσυνέλευση αυτή τη στιγμή είναι το μόνο δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο στη χώρα και εκείνοι έχουν καλέσει να ε, υπάρξει συνταγματικά απαιτούμενη ασυλία ε, για όλους τους βουλευτές, να γίνεται σεβαστή και να μην υπάρχουν άλλες διώξεις και καταστολές. Θα πρέπει να μπορούν την πολιτική τους θητεία, τις πολιτικές τους ευθύνες και το λειτουργήμά τους να το ασκούν χωρίς πιέσεις. Πριν καταφύγουμε σε βία για να επιλύσουμε την κατάσταση, θα πρέπει ε, να αποφύγουμε οποιαδήποτε ε, άλλη ενέργεια που θα προκαλέσει περαιτέρω παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πόνο και οδύνη στο λαό τη Βενεζουέλα. Ταυτόχρονα είναι σημαντικό να αποφύγουμε και την κλιμάκωση τη βία και τη εχθροπραξίε στη χώρα. Γι' αυτό ζητήσαμε να πάψουν οι εκφοβισμοί και οι επιθέσει στου πολιτικού εθνώντε και στου πολίτε και από τι διοκτικέ και από ένοπλε παραστατικέ δυνάμει. Θα πρέπει ο λαό τη Βενεζουέλας να μπορέσει επιτέλου να εκφράσει τη βούλησή του μέσω ελεύθερων προεδρικών εκλογών. Θα πρέπει να είναι ελεύθερε, αμερόληπτες δίκες, διαφανεί και να συμμετέχουν όλοι. Ε, είναι στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργηθεί μια διεθνής ομάδα επαφής για τη Βενεζουέλα, πράγμα που έγινε πρόσφατα. Σκοπός της λειτουργίας της ομάδας αυτής είναι να δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες για να ξεκινήσει πολιτική διαδικασία που θα οδηγήσει σε ελεύθερες και δίκαιες προεδρικές εκλογές. Η ομάδα επαφής έχει ορίσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για να εξακριβώσουμε κατά πόσο μπορούμε να, ενθαρρύνουμε να αποσπάσουμε εγγυήσει και να υπάρχει αξιοπιστία για τη δημοκρατική διαδικασία. Ε, τα σώματα, οι φορεί παρακολούθηση των εκλογών θα πρέπει να ξεκινήσουν ξεκινώντα από το εθνικό ε, εκλογικό ε, όργανο. Και επίση θα πρέπει να αλλάξει και ο εκλογικό νόμο. Όλα τα πολιτικά κόμματα και οι αρχηγοί του θα πρέπει να μπορούν να ανταγωνιστούν υποψήφοι ισότιμα. Οι πολιτικοί φυλακισμένοι πρέπει να απελευθερωθούν ανεξάρτητα τη πολιτική παρατήρηση θα πρέπει επίση να επιτραπεί στη χώρα. Η πρότασή μας δεν στοχεύει να δεσμεύσει κανένα να παρέμβει στα εσωτερικά της χώρας. Θα πρέπει όμως να υπάρξει μια διεθνής πρωτοβουλία για να υπάρχουν αυτές οι ελάχιστες προϋποθέσεις που εν τέλει θα οδηγήσουν στην ε, επανεκκίνηση μιας ε, λογικής δημοκρατικής διαδικασίας και την οργάνωση, διοργάνωση προεδρικών εκλογών. Επίσης πρέπει να δούμε και τις, ανάγκες, τις άμεσες ανάγκες του πληθυσμού. Δεν μπορούν να πληρώνουν το πολιτικό τμήμα της κρίσης ή ζωές τους απειλούνται. Η ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να μπορέσει να φτάσει στη χώρα χωρίς ε, φραγμούς και να φτάσει σε αυτούς που πάνω από όλα τη χρειάζονται. Τα τελευταία δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμεύσει πάνω από 67 εκατομμύρια ευρώ ανθρωπιστικής βοήθειας και ε, ανθρωπιστικής υποστήριξης και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε ακόμα παραπάνω. Ε, η ομάδα επαφή διερευνά τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα διεθνή μηχανισμό για τον συντονισμό και την παροχή ανθρωπιστική ε, συνδρομή στην Βενεζουέλα. Σε στενή συνεργασία με τον ΟΗΕ και τους διεθνείς και τοπικούς μας εταίρους. Θα πρέπει η βοήθεια να δίδεται αμερόληπτα βάσει των πραγματικών αναγκών του πληθυσμού και όχι βάσει των ε, πολιτικών προτεραιοτήτων και θα πρέπει να διανύμεται από ανεξάρτητους φορείς υπό την ηγεσία και την αιγίδα του ΟΗΕ η βοήθεια ποτέ δεν θα πρέπει να παίρνει πολιτικό χαρακτήρα. Θα πρέπει μόνο να αποσκοπεί σε ανθρωπιστικές ανάγκες και την κάλυψή τους. Η Διεθνής Ομάδα Επαφής εργάζεται αυτή τη στιγμή ε, εντατικά σε αυτούς τους δύο τομείς, τις εκλογές και την ανθρωπιστική συνδρομή και βοήθεια. Η ομάδα απέστειλε μια τεχνική επιτροπή για να διερευνήσει την κατάσταση στη Βενεζουέλα το Φεβρουάριο και να συζητήσει με όλε τι πλευρέ, τι προποθέσει και του όρου για να μπορέσουμε να οργανώσουμε αξιόπιστε και ανεξάρτητε προεδρικέ εκλογέ, αλλά και το τι θα γίνει με την ανθρωπιστική βοήθεια. Η ε, κυβερνητικοί υπεύθυνοι με του οποίου συζήτησε η ομάδα επαφή δώσαν κάποιε προτάσει, αλλά νέα ναι, προηγική συνάντηση θα γίνει και στα τέλη Μαρτίου κάπου στη Λατινική Αμερική. Εμεί οι Ευρωπαίοι δεν είμαστε ουδέτεροι. Πάνω από ένα εκατομμύριο Βενεζουελάνοι είτε έχουν πολιτικό διαβατήριο, είτε έχουν οικογένεια στην Ευρώπη. Μα νοιάζει ο λαό τη Βενεζουέλα. Μα νοιάζει αυτή η χώρα. Οι Βενεζουελάνοι ζητάνε αλλαγή και ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι η αλλαγή δεν μπορεί να επιβληθεί έξωθεν. Ε, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση διαρκεία, μια λύση μόνιμη, την οποία όμω να τη θέσουν σε εφαρμογή οι ίδιοι οι κάτοικοι τη χώρα. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα, ώστε ο λαό τη Βενεζουέλα να μπορέσει να διαφεντεύει την μοίρα του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα προχωρούμε στον κατάλογο των ομιλητών εκ μέρου των πολιτικών ομάδων. Πρώτο εκ μέρου του για δύο λεπτά, ο κύριο Κονθάλεφ Πόν. Κυρίε και κύριοι, αν σήμερα εμεί μέναμε χωρί ρεύμα, ε, σε μία ώρα όλοι οι ασθενείς που είναι στην εντατική θα πέθαναν. Ε, πέντε χρόνια θα μέναμε χωρίς ενσουλίνη, 20 ώρες, ε, δεν θα βγαίναν από τις βρύσες, δεν θα από τις βρύσες νερό. Θα χαλούσαν τα τρόφιμα που είναι στα ψυγεία σε μια μέρα. Σε δύο μέρες θα πέθαναν τα παιδιά που βρίσκονται στις θα πέθαιναν. Σε τρεις μέρες το αποθεκευμένο νερό δεν θα ήταν πλέον πόσιμο και από την πέμπτη μέρα και μετά θα πέθαναν οι ασθενείς που χρειάζονται μοκάθαρση. Αυτό θα ήταν μια μερα σε δυο μερες θα πέθαιναν τα παιδια που βρισκονται στις θερμοκοιτιδες σε τρεις μερες το αποθεκευμενο νερο δεν θα ηταν πλεον ποσιμο και απο την πεμπτη μερα και μετα θα πεθαναν οι ασθενεις που χρειαζονται μοκαθαρση αυτο θα ηταν μια τεράστια τραγωδία, μια τεράστια καταστροφή. Αυτό ακριβώ συμβαίνει στη Βενεζουέλα. Πάνω από 100 ώρε χωρί ρεύμα, χωρί ηλεκτροδότηση. Ο βενεζολάνικο λαό ε, είναι ανήμπορο εναντί στη φτώχεια, στην πείνα, τη δίψα, την έλλειψη φαρμάκων, στου εγκληματίε, ε, στι συμμορίε, ε, στην έλλειψη ενό εθνικού νομίσματο. Ο Νικολά Μαδούρο πλέον προσωποποιεί το θάνατο, το χάρο στη Βενεζουέλα. Και δεν μπορούν να λυθούν τα προβλήματα ε, από αυτούς που τα έλυσαν. Τα προβλήματα δεν μπορούν να τα λύσουν αυτοί που δεν τα βλέπουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιμείνει, πρέπει να απαιτεί την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων. Αρχές γενομένης από τον Λουίς Κάρλος Ντίαθ, έναν Ισπανό που αγνοείται γιατί έκανε τη δουλειά του, έκανε το δημοσιογραφικό του έργο. Θα πρέπει να αυξηθεί ο κατάλογος και ε, των ατόμων στους οποίους συμβάλλονται και την ε, λίστα των κυρώσεων. Δεν μπορεί να γίνονται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 εορταστικέ εκδηλώσει στη Μαδρίτη και να μην βλέπουμε τι τραβάει ο κόσμο εκεί. Πρέπει να στηρίξουμε το Γουαϊδό και την Εθνοσυνέλευση. Σήμερα βλέπουμε να κατεβαίνει στο ποτάμι το, ε, το πλήθο, το Καράκα, ε, για να πιει ε, νερό από το βόθρο. Η Βενεζουέλα είναι δημοκρατία, ελευθερία που ανήκει και σε εμά. Αν δεν το κάνουμε αυτό για τι πεπιθήσει μα, α το κάνουμε για τα 10 εκατομμύρια των Ευρωπαίων πολιτών που ε, είναι μαζί με το λαό της Βενεζουέλας, φυλακισμένοι του καθεστώτος. Ε, δεν θα αφήσουμε μόνο του ούτε τον Γκουαϊδό ούτε τον λαό της Βενεζουέλας. Ευχαριστώ. Και τώρα, λέω πρώτα εκ μέρους ομάδος S&D, το λόγο έχει ο κύριος Χουάρη Ατόντο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, δεν έχω λόγια για να καταδικάσω τον Μαδούρο. Ε, Παρ' όλα αυτά ε, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες πολύ δραματικές και σοβαρές εκτιμήσεις και λόγω της έλλειψης ηλεκτροδότησης, αλλά μακάρι να κάνω λάθος. Πιστεύω όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι η κίνδυνη μιας εσωτερικής σύγκρουσης στην Βενεζουέλα αυξάνονται. Είναι πιθανό να καταρρεύσει η χώρα. Αυτό θα δημιουργήσει μια κοινωνική τραγωδία ε, Χωρί λύση. Επομένω, κύριε και κύριοι, ομάδα επαφή. Ακριβώ γι' αυτό ε, είναι σωστή πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. για μια ειρηνική διαπραγμάτευση, ε, μια ειρηνική επίλυση τη σύγκρουση. και οι μόνοι που μπορούν σήμερα να συνομιλούν και με κυβέρνηση και με αντιπολίτευση είναι η της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ομάδα Κολυβία Κωνσταντίνα, Εκουαδόρη, η ομάδα επαφή αυτή. Αυτοί μπορεί να προωθήσουν την εσωτερική συμφιλίωση και ειρήνη. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε αντιμετωπίσουμε ε, την κοινωνική αυτή αντιπαράτευση μόνο με την ε, προσπάθεια για ειρήνευση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τάμπη για ένα λεπτό. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Πρόεδρε, η κατάρρευση του υδροελεκτρικού σταθμού ήταν άλλο ένα στερηπτικό κτύπημα κατά του λαού της Βενεζουέλας που έχει υποφέρει τόσα με ηθικό. Δύσκολο να εντοπιστούν τα αίτια λόγω των γελίων αιτιάσεων του καθεστώτος και των ΗΠΑ. Φαίνεται ότι μάλλον πρόκειται για την έλλειψη επενδύσεων και συντήρηση εξαιτία τη διαφθορά και τη κακοδιαχείριση του καθεστώτο. Και το οποίο συνεχίζεται τώρα. Όλε οι προσπάθειε επίλυση του προβλήματο επιδίνωσαν την κατάσταση και το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας εν γέννη υποφέρει και αυτό. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι υποφέρουν, τα νοσοκομεία δεν έχουν ρεύμα και απειλούνται και άλλες υποδομές. Καλό όλα τα κρατημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν πράξει να αναγνωρίσουν τον Γουαϊδό ως νόμιμο πρόεδρο της Βενεζουέλας ε, για να παράσχουμε κάποια ανακούφιση στον λαό της Βενεζουέλας. Να δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Βενεζουέλα ζει σε μια βαθιά κρίση μαζικών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, σπανίζουν τα τρόφιμα, τα φάρμακα, υπάρχει βία, καταστολή ε, πολιτική. Πάνω από τρία εκατομμύρια για αυτού τους λόγους εγκατέλειψαν ε, τη χώρα. Η στρατηγική κοινωνικού ελέγχου από το Μαδούρο μέσω της τιμωρίας και του εκφοβισμού είναι κάτι που μα προξενεί αποτροπιασμό και με θύματα πιο αδύναμους που υποτίθεται ότι θέλει να προασπίσει και τους ε, απειλεί και τελικά τους δόλοφων. Το λέει η Διεθνής Αμνηστία στην έκθεσή της της 20 Φεβρουαρίου. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Το 87% είναι στο κατόφλι της φτώχεια. Ο ελάχιστος μισθός είναι 6 δολάρια. Φυσικά είναι ελάχιστος με όλες τις έννοιες του όρου. Η Βενεζουέλα ε, είναι στη θέση 168 των πλέον διεφθαρμένων του κόσμου. Συρία, Σομαλία και Αφγανιστάν τη συνοδεύουν. Είναι χώρε που βρίσκονται σε πόλεμο γιατί ο Μαδούρο είναι σε πόλεμο με το λαό του όμως ε, τον ίδιο. Να μιλά κανείς ε, για δικαιοσύνη στην Βενεζουέλα είναι σαρκασμός, γιατί ο Μαδούρο ορίζει τους ε, δικαστές. Υπάρχει εκαθάριση από τη Βολιβαριανή Δημοκρατία. Το καταγγέλει η Διεθνή Αμνηστία στην έκθεση που σας προανέφερα. Και Πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες για βασανισμούς, για βασανιστήρια. Έχουμε την ε, ε, συνέλευση του Μαδούρο που σε καμία περίπτωση δεν κυβερνά ο νόμιμος πρόεδρος είναι ο Γουαϊδό. Πέντε μέρες έχει μείνει χωρίς ρεύμα. Παίρνει ο κόσμος ε, από τους υπονόμους, από τους οχετούς νερό για να πιει. Και η επανάσταση ε, θα γίνει από τους ε, Βενεζολάνους γιατί ζητούν τρόφιμα, ρεύμα, φως, ε, φάρμακα και τρόφιμα για τους αδελφούς μας από την Βενεζουέλα. Προσφέρω όλοι μας την αλληλεγγύη και για την κλεπτροκρατική τάξη του Μαδούρο θέλω να επιβληθούν κυρώσεις. Να μισή λεπτό, ο κύριος Κάουζο Περμούη τώρα, εκ μέρους της ομάδας Γκουεντζιέλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ζω ένα και δεν το λέω γιατί επανειλημμένως έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα της Βενεζουέλας αλλά γιατί επανειλημμένως το Κοινοβούλιο με πρόσχημα ε, την ανθρωπιστική βοήθεια ουσιαστικά έχει ε, κατά κάποιο τρόπο κλείσει τα μάτια μπροστά στις στρατιωτικές επεμβάσεις. Συρία, Λιβύη, τα ίδια ψέματα βλέπω. Δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα. Όταν το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να καταρρύψουν κυρίαρχες κυβερνήσεις ε, για να πάρουν το πετρέλαιο το φυσικό αέριο. Και τελικά θα έπρεπε ίσως να σκεφτούν ότι οδήγησαν στην πλήρη κατάρρευση ε, της Λιβύης, οδήγησαν στην κατάσταση που έχουμε σήμερα στη Ρία. Το ίδιο λένε και για τη Βενιζόλα, τα ίδια ψεύματα. Έχουμε τρομοκρατία στους δρόμους, μετά το πραξικό, μιλούν για ανθρωπιστική ε, κρίση, μιλούν για το ε, για τα blackout ως ένα πρόβλημα που είναι ένα πρόβλημα ε, διαχείρισης ε, και υπάρχουν ψεύματα για να βοηθήσουν τα ουσιέρα και στη Σουάνσικτον να προωθήσουν το χαρτί των Ηνωμένων Εθνών να καταρρίψουν, την ανατρέψουν την κυβέρνηση που δεν είναι του γούστου τους. Δεν τους ενδιαφέρουν τα 500 παιδιά που πέφτουν στη Γουαχέρα κάθε χρόνο ή τις δολοφονίες στην Κολομβία μέσα σε τρεις μήνες έχουν χάσει τόσοι άνθρωποι ε, στον κόσμο. Ε, βγάλτε τα χέρια σας, πάρτε τα χέρια σας μακριά από τη Βενεζουέλα και σταματήστε τα ψέματα. Ευχαριστώ. Κύριος Παπαδάκης, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, ένα λεπτό. Ε, παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι, κλείστε το μικρόφωνο. Γιατί θέλω να ακούσουμε τον κύριο Παπαδάκη, παρακαλώ, αγαπητέ. Συνάδελφοι, σας σας ακούσαμε. Ένα λεπτό κύριε Παπαδάκη. Ο λαό τη Βενεζουέλα είναι αρμόδιο να αποφασίσει ο ίδιο για το μέλλον του και για τι εσωτερικέ υποθέσει τη ίδια του τη χώρα. Καταδικάζουμε και καταγγέλουμε τα υπερελιστικά σχέδια που προωθούνται με προβοκάτσιε, ομάδε επαφή και όλα τα υπονομευτικά μέσα από τι Ηνωμένε Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι συμμαχικέ του κυβερνήσει στη Λατινική Αμερική για να ανατρέψουν τον εκλεγμένο πρόεδρο τη Βενεζουέλας βάζοντα τον αχυράνθρωπό του όλους αυτούς δεν τους πήρε ο πόνος για το λαό της βενεζουέλας. στο στόχαστρό του βρίσκονται ο έλεγχος της ενέργειας μιας πλούσιας σε πλουτοπαραγωγικές πηγές χώρας. καταδικάζουμε κάθε σενάριο για πραξικόπημα και υπερελιστική στρατιωτική επίδεση που βαφτίζεται ανθρωπιστική βοήθεια ή και άλλα προσχήματα. εκφράζουμε την αλληλεγγύη μα με το χτυπημένο από την καπιταλιστική κρίση λαό τη βενεζουέλας και τον αγώνα του κομμουνιστικού κόμματο βενεζουέλας. ο υπεριαλισμό δεν είναι ανίκητος. η πραγματική υπερδύναμη είναι η λαοί και αυτοί θα νικήσουν. Uh, uh, uh, Ευχαριστούμε για ένα λεπτό, κύριος Παντζέρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά το ψήφισμα που εγκρίναμε πριν από λίγες εβδομάδες στη τέλη Γενάρη, διερωτώμην, ποια είναι η βασική αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου και με ποιο τρόπο μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματο τη Βενεζουέλας. Το πρώτο νομίζω που θα έπρεπε να κάνουμε είναι να ξεχάσουμε τι διαθέσει προπαγάνδας και ε, χρησιμοποίησης ε, για ε, πολιτικού σκοπού στη συζήτηση αυτή. Πρέπει να ψάξουμε μια δημοκρατική διέξοδο από την κρίση αυτή με αξιόπιστε και ελεύθερε εκλογέ. Και να έχουμε επίγνωση ότι τη λύση που θα επιφέρουμε θα πρέπει να την επιφέρουμε δημοκρατικά και ειρηνικά. Δεν υπάρχουν άλλε επιλογέ θα δημιουργούσαν μεγαλύτερα προβλήματα και οδύνε για τον πληθυσμό. Είναι σημαντικό να φτάσει και ανθρωπιστική βοήθεια στη χώρα. Μόνο με κατάλληλε και νόμιμε οδού. Αυτέ είναι οι μόνε δύο επιλογέ και εναλλακτικέ που μπορεί να υποδείξει το Ευρωκοινοβούλιο. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν ε, προχειρότητα ή ευθυνότητα. Περιτή και επικίνδυνη αυτή τη στιγμή. Το μόνο που θα πρέπει να μα καθοδηγήσει αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είναι η πολιτική ευθεία. Ευχαριστούμε για 1,5 λεπτό η κυρία Μπεσέρα Μπαστερετσέα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε γιατί η Βενεζουέλα είναι στο σκοτάδι γιατί το χρειάζονται το σκοτάδι οι εγκληματίε για να διαπράττουν τα εγκλήματά του. Το καθεστώ του Μαδούρο είναι διεφθαρμένο, είναι ανίκανο. Γι' αυτό λοιπόν λείπει το φω και το τρόφιμα και τα φάρμακα από τη Βενεζουέλα. Είναι υπεύθυνο το καθεστώ του Μαδούρου για κάθε παιδί και για κάθε ασθενή που πεθαίνει λόγω του blackout σε ένα νοσοκομείο. Είναι επίση υπεύθυνο το καθεστώ για την παράνομη κράτηση του δημοσιογράφου Λουί Κάρλο Ντίεθ, που είναι ένα Ισπανό πολίτη, ένα Ευρωπαίο πολίτη. Το καθεστώ θέλει περισσότερο σκοτάδι για τα εγκλήματά του. Γιατί, Γιατί θέλει να ε, ε, εκτελέσει ε, χωρί να χρησιμοποιείται μία σφαίρα στο δυνατόν περισσότερους. Και γιατί θέλουμε αυτή τη διεθνή ομάδα επαφή, για να κάνει τον κλόουν, για να χάσει την αξιοπιστία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για πέντε μέρε. Τι κάνει αν δεν έχει ρεύμα, κλείνουν τα βενζινάδικα, δεν μπορεί να πάρει χρήματα, δεν μπορεί να πάρει νερό. Υπάρχει νόμιμο πρόεδρο στη Βενεζουέλα, έχει οδικό χάρτη. Είπαμε ότι θα τον πλαισιώσουμε, θα τον συνοδεύσουμε. Θέλουμε λοιπόν μεταβατική κυβέρνηση, θέλουμε εκλογέ. Και αν αυτό είναι το, έργο, αυτό είναι το πρόγραμμα του ΟΑΙΔΟ, αυτό θα το στηρίξουμε κι εμεί. Ε, και η κυρία Μογκερίνη, το μόνο που πρέπει να κάνει σε αυτή τη χώρα που είναι σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη είναι να ζητήσει ο πρόεδρο ΟΑΙΔΟ να τη πει τι ε, πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτόν και για του ε, Βενεζολάνου και να το κάνουν. Ευχαριστώ. Και τώρα για ένα λεπτό η κυρία Γκόμη. Let's see that χωρίς ηλεκτρικό ε, από αυτό εξαρτάται η ογεία για πολλούς. Χωρίς τρόφιμα, τα σχολεία κλείσαν, ε, παιδιά ε, γέροι αδύναμοι πληρώνουν τα κακανέα. Ο Μαδούρο πρέπει να διωχθεί από τη χώρα από τον ίδιο το λαό της Βενεζουέλας. Πρέπει να γίνουν ελεύθερες προεδρικές εκλογές. Θα πρέπει εξουσία να, περάσει στα χέρια του λαού. Δεν μπορεί να είναι στα χέρια μιας κλίκας γύρω από το Μαδούρο η εξουσία. Θα πρέπει να υπάρξει διεθνής δικαιοσύνη. Θα πρέπει το, οι κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Κούβας να καταλάβουν θα πληρήσουν ακριβά το τίμημα της καταστροφής ε, που προκαλεί η συμμορία του Μαδούρο ε, στη χώρα του. Ε, είναι θέμα χρόνου. Μόνο θέμα χρόνου. Δεν πρόκειται να διαρκέσει ο Μαδούρο στην κυβέρνηση, γιατί προκαλεί τεράστια οδύνη στο λαό τη Βενεζουέλα. Θα πρέπει ω προ αυτό να είναι απολύτω ξεκάθαρη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε και τώρα για 1,5 λεπτό η κυρία Χαράντσοβα. Ευχαριστούμε. Η Βενεζουέλα είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Τις τελευταίες ημέρες φάνηκε ότι είναι μία από τις βέβες ε, αποδείξεις ότι η χώρα δεν είναι αυτό που αξίζει η χώρα ως ηγέτης. Είναι ένας τύραννος κατάφορες παραβιάσεις και τα blackout είναι μια ακόμη απόδειξη του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παραμένει ε, σε κατάσταση αναμονής. Ε, θα πρέπει να επιβάλλουμε επιλεκτικές κυρώσεις. Θα πρέπει επίσης με ειρηνικό τρόπο η κυβέρνηση να εγκαταλείψει την εξουσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δύο επιλογές. Ε, να στηρίξει ενεργά μια νόμιμη ειρηνική και δημοκρατική λύση σαν αυτή που προτείνει ο Χουάν Γουαϊδό. Η δεύτερη επιλογή είναι να μείνει ε, στην αναμονή και να συνεχίσει ε, να γίνεται μάρτυρας δολοφονιών, ε, βασανιστήριων, πόνου και οδύνης. Μέχρι ότου καταρρεύσει πλήρως η Βενεζουέλα. Νομίζω ότι η επιλογή είναι στα χέρια μας και είναι σαφής. Πρέπει να σεβαστούμε τη δημοκρατία και το σύνταγμα της Βενεζουέλας και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τον Γουαϊδό ως προσωρινό πρόεδρος μεταβατικό Πρόεδρο. Ελπίζω σύντομα να δεχθούμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Πρόεδρο Γουαϊδό. Ευχαριστώ. Thank you. Έχω πολλά αιτήματα. Είμαστε όμω εκτό προγράμματο. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Να τηρήσετε παρακαλώ το ένα λεπτό όμω. Αλλιώ uh, κάποιοι δεν θα μιλήσουν. Αναγκαστικά. Γαλάζια κάρτα. Όχι, είστε στον κατάλογο των μιλητών. Ε, ε πολύ αργά. Λυπάμαι. Ε, έχετε τον λόγο πάντως, είστε πρώτος στον κατάλογο. Πρόεδρε, η κατάσταση στη Βενεζουέλα είναι κατάσταση που έχει ξεφύγει από τον έλεγχο. Δεν υπάρχει ηλεκτρικό η κατάσταση είναι κατάσταση απελπισίας και πείνας. Χρειάζεται απελπισμένα ε, ο κόσμος νερό, ε, τα νοσοκομεία, η κλινική υποστήριξη, η υγειονομική περίθαλψη, οι ζωές των ανθρώπων κινδυνεύουν. Αυτό δεν είναι πλέον πρόβλημα απλώς δικτορίας ή δημοκρατίας. Είναι θέμα ζωής ή θανάτου είναι πρόβλημα ανθρωπιστικής κατεπίγουσας ανάγκης. Πρέπει να πούμε εδώ ότι πολλές φορές αυτό το κοινοβούλιο πολλοί βουλευτές κατήγγυλαν ε, ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Και αυτό είναι υπέρ τους, διότι εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η υπόλοιπη διεθνής κοινότητα, δεν αναγνωρίσαμε εγκαίρως ότι ο Μαδούρο είναι δικτάτορ. Και όχι απλώς είναι δικτάτορ, είναι τύρανος τύρανος ο οποίος κάποια στιγμή θα πρέπει να θεωρηθεί και ε, δολοφόνος του λαού του. Ευχαριστούμε, αλλά θα πρέπει να παραμείνουμε στον του κύριε Ρανζέλη, γιατί έχουμε πολύ μακροσχελή κατάλογο και δεν θέλω να κλέψω χρόνο από κανέναν. Ο κύριος Φαρία για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο αγώνα μου για την ελευθερία και τη δημοκρατία στην Βενεζουέλα δεν είναι σημερινή όπω συνέβη με κάποιου συναδέλφου που τώρα ανακάλυψαν το θέμα. Γι' αυτό θα θέλαμε η Βενεζουέλα να μην καταλήξει έτσι. Είναι τραγικέ οι συνέπειε. Είναι ε, απελπιστική κατάσταση με τα τρόφιμα και τα νοσοκομεία. Τα μωρά και οι άρρωστοι πεθαίνουν εξαιτία τη δικτατορία του Μαδούρου. Το καθεστώ του Μαδούρου είναι υπεύθυνο για την κατάσταση του ηλεκτρικού συστήματο τη χώρα και των οικονομικών κυρώσεων των ΗΠΑ που έχουν επιβληθεί στη χώρα. Γι' αυτό φεύγουν και διαφεύγουν από τη χώρα εκατομμύρια πολίτε. Ε, το πρόσφατο ηλεκτρικό βρακύκλωμα είναι αποτέλεσμα τη ανευθυνότητα ενό δικτατορικού καθεστώτο που έκανε ό,τι μπορούσε για να στείλει χρήματα, πετροδολάρια που παράγονται στη χώρα προς ε, πολλές εταιρείες offshore. Αυτές ε, οι ε, κλεπτοκάρτες που έχει χρησιμοποιήσει η Βενεζουέλα μέσω του στρατιωτικού της συστήματος θα πρέπει να σταματήσουν να χρηματοδοτούν αυτές οι εγκληματικές δραστηριότητες. Ευχαριστούμε. Η κατάσταση στη Βενεζουέλα είναι δραματική. Είναι τραγική. Ε, και απειλούνται οι ζωές μητέρων, ε, ε, μωρών, ολόκληρων οικογενειών. Θα πρέπει να πω ότι με τις απόψεις που ακούστηκαν εδώ στην Ολομέλεια πρέπει να πούμε ότι κάποιες από αυτές δεν είναι ρεαλιστικές, ούτε απηχούν το τι πραγματικά συμβαίνει στη χώρα. Η πολιτική μας παρέμβαση θα πρέπει να είναι πολύ στοχευμένη και περιορισμένη. Θα πρέπει να κοιτάξουμε, να κινητοποιήσουμε τη διεθνή κοινή γνώμη και να αποστείλουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Το σημαντικότερο είναι η Βενεζουέλα να υποστηριχθεί στα σημερινά της προβλήματα. Η χώρα αυτή έχει προβλήματα από το 1948 Τώρα αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε είναι να παρακολουθούμε την κατάσταση και να αποστέλουμε ανθρωπιστική βοήθεια και κάτι παραπάνω. Ευχαριστούμε κύριο Σαλαφράγκα Σάντζερ για ένα λεπτό η κυβέρνηση παραμένει ε, στην εξουσία, αγκιστρώνεται στην εξουσία μόνο με τη βίαιη άσκηση ε, ισχύω ε, σε βάρος του πληθυσμού της. Πόσο ακόμα πρέπει να υποφέρει, είναι η ερώτηση, η κοινωνία. Πόσοι ακόμη πρέπει να πεθάνουν στο σοσιαλιστικό πείραμα του 21ου αιώνα μέχρι να οδηγηθεί σε οριστική κατάρρευση. Η χώρα βρίσκεται σε μια πλήρως χαοτική κατάσταση, κύριε Πρόεδρε. Ωστόσο, η κατάσταση καταστολή δεν σταματά. Θέλω και εγώ να αναφέρω στον δημοσιογράφο που ανέφεραν οι προλαλήσαντε, που ζητάμε την άμεση απελευθέρωσή του Είδαμε τι έγινε με το πλήρωμα της Air Europa. Είδαμε ότι καταστρέφεται η ανθρωπιστική βοήθεια στα σύνορα με Βραζιλία και Κολομβία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί όμως να παραμένει απαθήσα μπροστά σε αυτές τις κατάφορες συστηματικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να αυξηθούν οι κυρώσεις και κύριε Επίτροπε πράγματι οι διπλωματικές κυρώσεις πρέπει να εφαρμοστούν. Δεν άκουσα ούτε μία διαμαρτυρία Διακόπτεται ο μιλητή για ένα λεπτό, κυρία Χιμένεθ. Μία από τις πιο πλούσιες ε, ε, φυσικούς πόρους ε, χώρες έχει μείνει χωρίς ρεύμα πέντε μέρες και ζει τη χειρότερη χρήση της ιστορίας του και γι' αυτό δεν φταίνει ε, ρεπουμπλικανοί και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος, αλλά το σοσιαλιστικό πείραμα ε, στη Βενεζουέλα, οι πολίτες όπως είπαν και οι συνάδελφοί μου ε, πάνε να πιούν μολυσμένο νερό, πεθαίνουν παιδιά στα νοσοκομεία. Από το 2013 όμως οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στη Βενεζουέλα έχουν στρατιωτικοποιηθεί από ό,τι φαίνεται και η Κούβα συνεχίζει να παίρνει 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο σαν βαμπύρ ε, να ε, τα παίρνει από τη χώρα αυτή. Και όλα αυτά πλήττουν το λαό της Βενεζουέλας. Έχουμε το μεταβατικό πρόεδρο ε, Γουαϊδό ε, και στέλνονται κατά προτεραιότητα αυτά τα ε, βαρέλια πετρέλαιο στην Κούβα όλο αυτό τον καιρό. Ε, αυτά είναι τα πράγματα που πρέπει να αποφασίσουμε. Επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. πίνα, έλλειψη φαρμάκων, διαφθορά ε, κάνουν ασφικτιά ε, η χώρα της Βενεζουέλας εδώ και χρόνια. Έχασε τις εκλογές ε, ο Μαδούρο, αλλά εφήβρε τη λύση της Εθνοσυνέλευσης. Μετά είχαμε το, τα blackout που δείχνουν πόσο ανίκανη είναι αυτή η κυβέρνηση, είναι αυτό το καθεστώς. Ήδη τον ερευνούν και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ορισμένοι διεθνείς οργανισμοί, λέει κυρία Μπιλμπάου Μπαραντικά. Ακούσαμε θύματα του Μαδούρο, ακούσαμε ανθρώπους με μόρφωση που θα είχαν μέλλον αν ζούσαν οπουδήποτε αλλού. Άντρε και γυναίκε καταδικασμένοι στη φτώχεια, στην περιθωριοποίηση, που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια, την οποία μπλοκάρει ο δικτάτορα. Θέλουν μια χώρα ελεύθερη, μια χώρα ε, ειρηνική. Και η λύση περνάει από αυτή την ομάδα επαφή για μια κοινή λύση για τη διοργάνωση αξιόπιστων ελεύθερων εκλογών. Θέλω να εκφράσω την αντίθεσή μου σε οποιαδήποτε λύση ε, που δεν θα γίνει ε, στο πλαίσιο του διεθνού δικαίου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μιράντα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Blackout. Ναι, πράγματι υπάρχει ένα blackout, αλλά όχι μόνο σε ό,τι αφορά την εκδοδότηση, αλλά και σε ό,τι αφορά την πληροφόρηση. Δεν βλέπουμε και τα δύο πραγματικότητες. Δεν ξέρω αν είδατε, κύριε Επίτροπε, το άρθρο ε, των New York Times. Δεν νομίζω ότι είναι ε, συνένοχη του Μαδουρό. Όμω, πολλά ψευδέ ιστορίε και μύθου ε, του καταρρύπτει αυτό το δημοσίευμα και πολλοί ε, συντηρητικοί βουλευτέ φαίνεται να μην ενδιαφέρονται τελικά τόσο για τη Βενεζουέλα, αλλά κάνουν ε, λόγου για εσωτερική ισπανική κατανάλωση για να ξαναβγούν σε εκλογέ. Ούτε του ενδιαφέρει η ομάδα επαφή του Μοντεβιδέο. Τον μποϊκοτάρουν συνεχώ, ενώ αυτό προσπαθεί να βρει λύση βασισμένη στο διάλογο. Και επειδή μιλάμε για διάλογο, αν εσεί δεν θέλετε διάλογο, αλλά business as usual, αν θέλετε business, πετρέλαιο, χρήμα, χρήμα και χρήμα, θα πρέπει να ανησυχήσετε. Θα πρέπει να ανησυχήσετε γιατί τρίζει η καρέκλα σα. Ε, και αυτοί που θα έχουν τις έδρε σα σύντομα θα είναι οι ακροδεξοί. Και αυτό θα πρέπει να σας ανησυχεί. Ευχαριστώ. Σένρα για ένα λεπτό. Sí. Gracias, Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, τέσσερα πράγματα θα σα ζητήσω. Κύριε Επίτροπε, να αφήσετε την Βενεζουέλα ήσυχη. Πρώτον, όπω είπε ο Επίτροπο, οι Βενεζολάνοι, άντρε και γυναίκε, είναι αυτοί που αποφασίζουν για το μέλλον του. Δεύτερον, μην είστε κοινικοί αν πράγματι σα ενδιαφέρει η δημοκρατία, αν σα ενδιαφέρουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, να καταδικάσετε ε, τι εγκληματικέ ενέργειε και τις κυρώσεις ε, των ΗΠΑ. Επιθέσεις όπως αυτές ε, που δημιούργησαν τα blackout. Δεν μα λένε από πού προέρχονται αυτά τα blackout. Τρίτον, να δείξετε ότι σα ενδιαφέρει ο λαό τη Βενεζουέλα και όχι το πετρέλαιο τη χώρα Και τέταρτον, να πάρτε τα χέρια σα από τη Βενεζουέλα και χρησιμοποιήστε το χρόνο σα για να καταρτήσετε πολιτικέ που πραγματικά θα τερματίσουν πλουτίσουν τη φτώχεια τη εργατικής τάξης ε, και δεν θα κάνουν να πλουτίσουν περισσότερο πολυεθνικέ. Ευχαριστώ. Πιμέντα λόπε για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Βλέπουμε ότι στις συζητήσει για τη Βενεζουέλα εδώ δεν υπάρχει καμία ειλικρίνεια. Διαρκώς ψευδόμεθα χωρίς καμία, κανένα όνειδος. Θα πρέπει να ζητήσουμε από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να ε, να αναλάβει απλώς ευθύνε, αλλά όχι υπό την πίεση τρομοκρατικής ε, πίεσης, όπως ξέρουμε ότι έγινε με την απόπειρα πραξικοπίσματος. Διαρκώς ακολουθείτε την κυβέρνηση Τραμπ και αφήνετε τα πράγματα να πάρουν τον δρόμο τους, αλλά αυτό έχει οδηγήσει σε παταγώδη επιτυχία. Παταγώδη επιτυχία στα σύνορα, παταγώδη επιτυχία στον ηλεκτροδότηση της χώρας, παταγώδη επιτυχία στην οικονομία. Ε, επιτυχία. αποτυχία. Εδώ λοιπόν πρέπει να βοηθήσουμε τη χώρα και να προωθήσουμε τις κοινότητες που μπορούν να υποστηρίξουν τη χώρα και να την οδηγήσουν στο δρόμο της νομιμότητας. Δεν θα πρέπει να, ε, πιε, να καταστέλουμε τη δράση ενός λαού που βασίζεται στην παράδοση του Μπολιβάρ. Ευχαριστούμε. Thank you. Ευχαριστώ. Η κατάσταση στη Βενεζουέλα είναι μια απόλυτη τραγωδία. Εκεί μας πήγε ο σοσιαλισμός που κάθε φορά που αναλαμβάνει την διακυβέρνηση μιας χώρας οδηγεί στην καταστροφή. Απόλυτο σοσιαλισμό απόλυτη καταστροφή. Ο λαό τη Βενεζουέλα ζει μια ανίποτη τραγωδία. Και το μόνο που θα μπορούσα να πω ότι κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα είναι οι απόπειρε παρέμβαση. Θα έλεγα η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι διεθνεί παίκτε να είναι πολύ προσεκτικοί όταν προσπαθούν να επέμβουν δημοκρατικά για να βοηθήσουν, διπλωματικά με συγχωρείτε, για να βοηθήσουν το λαό της Βενεζουέλας. Κύριε Πίτροπε, νομίζω ήρθε η σειρά σας. Παρακαλώ. This has been a very useful... Η συζήτηση ήταν πολύ χρήσιμη. Ευχαριστώ τους κυρίους και τις κυρίες βουλευτές για τις παρεμβάσεις τους. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Βενεζουέλα θα συνεχίσει να συμπεριλαμβάνει τόσο πίεση όσο και πολιτική συμβολή στην εξασφάλιση μιας δημοκρατικής ειρηνικής λύσης. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις χώρες της περιοχής και με άλλους διεθνείς παίκτες, κυρίως μέσω της Διεθνούς Ομάδας Επαφής και να αξιοποιούμε οτιδήποτε έχουμε στη διάθεσή μας για να οδηγηθεί η χώρα σε μια ειρηνική λύση μέσω διαπραγματεύσεων. Η βασική μας ανησυχία είναι η κατάσταση του λαού της Βενεζουέλα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε τις δικέ του ανάγκες κατά πρώτο λόγο και να πω εγκατακλείδη ότι εκτιμώ βαθύτατα τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο διατηρεί το θέμα αυτό υψηλά στην διεθνή ατζέντα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, Ένα συνάδελφος ζήτησε τον λόγο στο πλαίσιο του Catch και δυστυχώ ε, ενημερώθηκα ενώ είχαμε ήδη ξεκινήσει. Όταν κλείσει ο κατάλογο των μιλητών, Δυστυχώ ε, κλείνει, συγγνώμη, λυπάμαι πραγματικά, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Ευχαριστώ. All μικρόφωνο. down Μίλησε στο μικρόφωνο, παρακαλώ. Ε, όλο εκτάκτο κάνω μια εξαίρεση. Παρακαλώ, μιλήστε από τη θέση σα. Δεν θέλετε το λεπτό. Όχι, θα μιλήσω, θα μιλήσω. Λέει ο βουλευτή. Γρήγορα, παρακαλώ. Εν πάση περιπτώσει, υπενθυμίζω τον κανόνα. Όταν κλείνει ο κατάλογο των μιλητών στο Catch the και ζητήσετε μετά τον λόγο, μπορεί να λάβετε τον λόγο. Αλλά υπάρχουν όρια. Επειδή δεν είδα τη συνάδελφο, γι' αυτό κατ' εξαίρεση τη δίνω το λόγο για ένα λεπτό, παρακαλώ. Θα μιλήσω από εδώ. Η Βενεζουέλα ζει στο σκοτάδι τώρα, αλλά το ξέραμε και από πριν. Ε, υπάρχει μια ανευπροηγουμένη ανθρωπιστική κρίση ε, που είναι στη μεταφορικά ε, μια κατάσταση στο σκοτάδι. Τώρα όμως είναι και κυριολεκτικά στο σκοτάδι χώρα. Παιδιά που ζουν ε, ε, χωρίς ρεύμα και κινδυνεύουν. Είδαμε τι έκανε στα σύνορα ο Μαδούρο που έστελνε πίσω τα φορτηγά που έκαιγε ε, τα φάρμακα για τους ασθενείς, έκαιγε τα τρόφιμα για τους πεινασμένους. Ε, ε, θέλουμε την ομάδα επαφής, θέλουμε το διάλογο. Όμως εδώ και μήνες και χρόνια δεν κάνει τίποτα η Βενεζουέλα. Πώς θα μιλάμε για ελεύθερες εκλογέ έτσι στον αέρα. Πρέπει να συνομιλούμε με τον Γουαϊδό και να μας πει συγκεκριμένα τι θα κάνει ο Μαδούρο. Ποτέ δεν πρόκειται να συγκαλεί σε ελεύθερες εκλογές. αυτό που θέλω να πω στο γενναίο λαό διακόπτεται. Η ομιλητρία. Το ίδιο ε, ισχύουν για όλους. Ένα λεπτό ήταν ε, ο χρόνο που είχατε στη θέση σα και παραλαμβάνω τον κανόνα για την διαδικασία κατηδία. Τέλο πάντων, εδώ ολοκληρώθηκε η συζήτηση και θα ψηφίσουμε στην προσεχή συνδολομέλεια και περνάμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη που είναι η έκθεση τη κυρία Φωτίγκα. Συνέχεια που έχει δώσει η ΕΕ στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση τη προπαγάνδα εναντίον τη από τρίτου. Κύριε Σιγήτρια, κύριε Φωτίγκα, έχετε τέσσερα λεπτά. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, έχω την τιμή να παρουσιάζω τις συστάσεις προς το Συμβούλιο και την υπατή εκπρόσωπο για τα θέματα εξωτερική πολιτικής. Τέσσερα χρόνια μετά από την υιοθέτηση, την έγκριση της μαρικής έκθεσης για την Stratcom τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για την αντιμετώπιση δηλαδή της εχθρική προπαγάνδας κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτα μέρη. Ήμουν εισηγήτρια για την άλλη έκθεση επίσης. Θέλω να υπενθυμίσω ότι η πρώτη έκθεση εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2016. Είχε δύο μέρη που αναφέρονταν στους βασικούς πρωταγωνιστές, στους βασικούς παίκτες αν θέλετε, στην προσπάθεια αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει την εχθρική προπαγάνδα από τρίτα μέρη. Πρόκειται για κράτη, την Ρωσική Ομοσπονδία κατά κύριο λόγο, αλλά και για μη κρατικού φορεί, κυρίω ριζοσπαστικοποιημένου φορεί όπω ο ΕΣΥΣ. Αυτή τη φορά οργανώσαμε λίγο καλύτερα τις συστάσει μα, με τρόπο εν τέλει διαφορετικό χάρη στι συνεισφορέ από διάφορε πολιτικέ ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι, διαχωρίσαμε την έκθεση πρώτον στην κατάσταση το 18. Αναφερόμαστε στον ευρύδικο πόλεμο που αντιμετωπίζουμε. Τονίζουμε εν συνεχεία την αναγκαιότητα να αποφύγουμε τη λογοκρισία στην προσπάθεια αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης και των ψευδοειδήσεων. αυτές τις στάσεις που βάλουμε στα κράτη-μέλη και στο Συμβούλιο. Τονίζουμε την αναγκαιότητα ποιοτική δημοσιογραφίας, την σημασία της ελευθερίας του λόγου και των μέσων. Επίσης, τονίζουμε την δυνατότητα λήψης νομοθετικών μέτρων ή κανονιστικών μέτρων σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ακόμα και στο ανθρωπιστικό δίκαιο θα μπορούσαμε να θεσπίσουμε μέτρα